Και περνάμε στο πρώτο σημείο της ημέρησης διάταξης που είναι η δήλωση του Συμβουλίου καθώς και της Κομισιόν για τα μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων του ρεύματος μετανάστευσης που προέκυψε από τον πόλεμο της Συρίας. Δίνω καταρχήν το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, τον κύριο Λεσκοβίτσιους. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Κατά τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλά σημαντικά γεγονότα στην Συρία, τραγικά γεγονότα, αλλά τώρα η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Ο αριθμός των προσφύγων που έχουν καταγραφεί, περιμένουν να καταγραφούν, ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Πάνω από του Μισού είναι παιδιά, ένα τέταρτο είναι γυναίκε και παραπάνω. Όπως ε, βρισκόμαστε εδώ και συζητούμε, συνεχίζει να διωγγώνεται το μεταναστευτικό ρεύμα από την Συρία. Τα άτομα αυτά που είναι πρόσφυγες έχουν περάσει στιγμές και γεγονότα βίας και έχουν εκτοπιστεί από τις αιστείες τους. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους ε, γείτονες της ε, Σουρίας, Συρίας. Σε ό,τι αφορά τους εσωτερικά εκτοπισμένους μέσα στη Συρία, ο ΙΕ εκτιμά ότι μπορεί να φτάσουν τα 3,5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλοί Σύριοι οι οποίοι κινούνται προς τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το Συμβούλιο παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τα προβλήματα που προκύπτουν από το μεταναστευτικό αυτό ρεύμα ε, πολιτών της Συρίας. Το θέμα αυτό συζητήθηκε χθες στο Συμβούλιο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης στο Λουξεμβούργο και σε αυτή τη συνάντηση τόνισε και πάλι η Υπουργή την απόλυτη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την αρρωγή που δίδεται στους πρόσφυγες αυτούς λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Κομισιόν και τα αποτελέσματα μιας διερευνητικής αποστολής για τα θέματα των προσφύγων της Συρίας. Γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι η κλίμακα αυτού του δράματος, που είναι και ένα τεράστιο βάρος για τις κυβερνήσεις των ομόρων χωρών, όπως είναι η Ιορδανία, η Τουρκία, το Ιράκ κτλ. Εμεί θέλουμε να επενέσουμε τους γείτονε τη Συρίας για το γεγονός ότι κράτησαν τα σύνορά του ανοιχτά. Και ενθαρρύνουμε τι χώρε αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Από την άλλη μεριά η διεθνής κοινότητα έχει απόλυτη ευθύνη να συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη σε αυτούς οι οποίοι γενναιόδωρα έχουν υποδεχθεί ένα μεγάλο μέρο. ε, προσφύγων. Έχουμε σταθεί στο προσκήνιο λοιπόν της παροχής βοήθειας σε όλους αυτούς τους πρόσφυγες. Κάθε κράτος μέλος προσπαθεί να βρει τρόπους για να καταπραίνει τα βάσανα των σύρων προσφύγων και στη χώρα τους και έξω από τη χώρα τους. Παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα και τους περιορισμούς στον προϋπολογισμό. Ξεπερνάει το 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση για τα ανθρωπιστικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά 412 εκατομμύρια έχουν δοθεί σε διάφορα ανθρωπιστικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων αυτών που μπορούν να επωφεληθούν. Είναι σχεδόν λοιπόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, βοήθεια προς τους πρόσφυγες. Με τον τρόπο αυτό ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι πρόσφυγες την χάνουν υποστήριξης και υπάρχει απόλυτη ε, λογοδοσία από την πλευρά των δικών μας αρχών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν προοπτικές για μια ε, άμεση λήξη των εχθροπρασιών στην ε, Συρία. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει και μέτρα τα οποία μπορεί να είναι μέσω πρόθεσμα και, και μακροπρόθεσμα. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο δηλαδή, να υποστηρίξουμε τους πρόσφυγες, αλλά να εξασφαλίσουμε την ανοικοδόμηση των τοπικών κοινοτήτων στη Συρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με διεθνούς εταίρους προετοιμάζει ένα πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο σαν στόχο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από την κρίση Ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα του χρόνου. Το Συμβούλιο χαιρέτησε την ε, πρόοδο για την επίτευξη αυτού του προγράμματος και προσκάλεσε την Κομισιόν να συνεχίσει τις προσπάθειές της για αυτό το τόσο σημαντικό έργο. Η επανεγκατάσταση των σύρων προσφύγων οι οποίοι χρειάζονται προστασία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα μοναχά από τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει μας υπόψη και εξετάζουμε. Αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους πρόσφυγες και αυτό το θέμα είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως γνωρίζετε, και του Συμβουλίου, που συνεχίζονται. Πρόεδρε, μέλη της Κομισιόν, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιμετωπίζουμε σήμερα ένα ιδιαίτερο θέμα με το μεταναστευτικό ρεύμα των προσφύγων. Δεν πρέπει όμως να ξεχάσουμε τον πιο σημαντικό στόχο μας να μπορέσει να σταματήσει αυτή η σύγκρουση και να προχωρήσουμε προς μια πραγματικά δημοκρατική Σύρια. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου υπογραμμίσαμε την ανάγκη για μια πολιτική λύση και την ανάγκη να υπάρξει δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας για να μπορέσει να προωθήσει την ειρήνη. Η ύπατη εκπρόσωπος έχει χαιρετήσει την, το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία ως ένα κέριο βήμα προς την επίτευξη μιας βιώσιμης και μόνιμης λύσης στην κρίση της Συρίας. Ακολουθεί αυτό μια πολύ σημαντική ε, μια σημαντική <clears throat> απόφαση που ελήφθη από το Συμβούλιο του ΟΣΑ στην Χάγη. Υπάρχει επίσης και ο κίνδυνος που προέρχεται από όπλα μαζικής καταστροφής. Εδώ το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρξει απόλυτη λογοδοσία σε σχέση με τα όπλα αυτά και θα πρέπει να υπάρξει μια στεναρή διεθνής αντίθεση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονίσει πάντα ότι είναι έτοιμη να υποστηρίξει όλες τις δράσεις που προβλέπονται από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και ε, υποστηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου για τα όπλα μαζικής καταστροφής της Χάγης. Πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε με αυτήν την ε, ορμή που έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία, τα Ηνωμένα Έθνη, τα Αραβικά κράτη, όλοι πρέπει να συνεργαστούν για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια διεθνή λύση βιώσιμη και το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει <clears throat> τονίσει ότι μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τη συμφωνία την προσωρινή της γενέβη του 2011 και ζητά να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στο ταχύτερο δυνατό. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα τελευταία δύο χρόνια η κατάσταση στη Συρία έχει επιδεινωθεί και είναι πια ένας πλήρης εμφύλιος πόλεμος, του οποίου τα κύρια θύματα είναι οι άμαχοι στη Συρία είναι μεγαλύτερη παραποτέ η ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη έχουν κάνει εξαιρετικέ συμβολές στο να υπάρξει αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια και θα είναι πάντα στην πρωτοπορία των προσπαθειών για να εξασφαλιστεί αυτή η βοήθεια και φυσικά εμείς πρέπει να συγκεντρώσουμε καλύτερα τους πόρους μας και να έχουμε μια αποτελεσματική βοήθεια στον τομέα αυτό. Το Συμβούλιο καταγράφει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά που καταδεικνύει και πάλι το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παρακολουθήσει με μεγάλη προσοχή το θέμα αυτό και τις πιθανές επιπτώσεις αυτής της σύραξης στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως, μια ανθρωπιστική πολιτική είναι απαραίτητη και είναι ε, πρωτεύω να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα συντονισμένης δράσης και χρήσης της δράσης των κρατών μελών και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Ε, τη δήλωση της Επιτροπής θα κάνει σήμερα ο Επίτροπος κ. Μπαρνιέ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές που πάλατε τη συζήτηση αυτή στην εμερήσια διάταξη. Μια κατεπίγουσα συζήτηση για ένα πολύ σοβαρό, τραγικό μάλιστα φαινόμενο. Η Σεσίλια Μάστρομ είναι μαζί με τον κύριο Μπαρόζο στη Λαπετούσα. Άλλοι συνάδελφοι είναι στις Ηνωμένε Πολιτείε. Εκ μέρους τους λοιπόν εγώ θα σας παρουσιάσω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα που ακούσαμε τον ε, Λιθωνό Αντιπρόεδρο. Τα πρώτα μου λόγια έρχονται μετά από το ένα λεπτό σιγή που είχε χτες το Κοινοβούλιο ως εκδήλωση αλληλεγγύης προς όλα τα θύματα, τις οικογένειές τους, μετά τη νέα αυτή τραγωδία που είχαμε στη Λαμπεντούσα πριν από μερικές μέρες. Με τόσα θύματα. άντρες, γυναίκες, παιδιά που προσπαθούσαν να δραπετεύσουν από την σύραξη στην ε, Μέση Ανατολή ή από την Αφρική. Οι διεθνείς πρωτοβουλίες κυρίες και κύριοι και ιδιαίτερα η Ρωσοαμερικανική Συμφωνία για τον έλεγχο και την καταστροφή των χημικών ε, όπλων στη Συρία που είναι υπαρκτό. Το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών έχει σαν αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί η πιθανότητα στρατιωτικής απάντησης από πλευράς των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κατάσταση στη Συρία σταθεροποιείται. Αντίθετα, οι στρατιωτικές δραστηριότητες συνεχίζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της είπα της εκπροσώπου, της συναδέλφου μας Κάθη Άστον, υπογράμμισε την ανάγκη κατεπηγόντως για μια πολιτική λύση. Είναι ο μόνος δρόμος για να σταματήσει ο πόλεμος αυτός και επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να δράσει και να δώσει τέλος στη σύραξη αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επαναλάβει ότι είναι στην διάθεση των διαφερμένων μερών να βοηθήσει και στα πλαίσια του Συμβουλίου του ΙΑΚ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε επαφή με το ΙΑΚ προκειμένου να δει πώς μπορεί καλύτερα να βοηθήσει επιτόπου. Στη σύραξη αυτή, ή κάτι άστον έτσι σκέφτεται πάντως, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα που έχει η στιγμή αυτή ολόκληρη η διεθνής κοινότητα. Γι' αυτό και εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους μας τους εταίρους και τις Ηνωμένε Πολιτείε, εννοείται, αλλά και με τη Ρωσία, τις αραβικές χώρες, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια πολιτική λύση από πλευρά της διεθνούς κοινότητας που να είναι μια λύση με μια φωνή. Το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας επικυρώνει την συμφωνία της 30 Ιουνίου του 2012 που λέει ότι όσο γίνεται πιο γρήγορα πρέπει να προχωρήσουμε σε λύση. Και όπως λέει ξεκάθαρα εδώ ο Αντιπρόεδρος, είμαστε αντιμέτωποι με μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς κρίσεις. Διότι εδώ ένα τρίτο του πληθυσμού της Συρίας ουσιαστικά μετατοπίζεται, δύο εκατομμύρια έχουν καταγραφεί ήδη από την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, έχουν μετακινηθεί προς τις γείτονες χώρες δηλαδή, και ο Λίβανος και η Ορδανία που γνωρίζω, ε, η Τουρκία, η Αίγυπτος δέχονται επίση πρόσφυγες. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης θέλω να υπογραμμίσω ότι αρχές της χώρες αυτές δεσμεύτηκαν να δείξουν αλληλεγγύη απέναντι στους Σύριους πρόσφυγες. Η ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών εκτιμάει ότι μέχρι τα τέλη της χρονιάς αυτής οι Σύριοι πρόσφυγες σε ολόκληρη την περιοχή, στις γείτονες χώρες δηλαδή με τη Συρία, θα φτάσει στα 3 ή στα 3,5 εκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα βρίσκεται και βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή της διεθνούς βοήθειας απέναντι στους πρόσφυγες αυτούς. δύο δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη δοθεί από τα τέλη του 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη υπό τον έλεγχο βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να στηρίξουμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος δωρητής με διαφορά στην κρίση αυτή. Αλλά και εμείς φτάνουμε σε κάποια όρια το 2013. Θέλω επίση εδώ να διευκρινίσω ότι 56% της ανθρωπιστικής αυτής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών ε, απευθύνονται στις γείτονες χώρες προς τη Συρία. 44% πηγαίνει στην ίδια τη Συρία. Μέσω διαφορών οργανώσεων εκεί. Οι γείτονες χώρες, ο Λίβανος και η Ιορδανία, κατά πρώτο λόγο, Υπογραμμίζουν επίσης ότι οι δυνατότητες που έχουν για να βοηθήσουν φτάνουν στα ωριά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη μεριά κάνει ό,τι μπορεί ώστε οι Σύριοι πρόσφυγες σε όλες αυτές τις γείτονες χώρες όπου καταλήγουν να έχουν ε, αρκετή ανθρωπιστική βοήθεια και νομική προστασία. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, Υπάρχει ένα πρόγραμμα περιφερειακής προστασίας που συμπληρώνει τα πρώτα προγράμματα που είναι βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ολοκληρώνεται τώρα σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τους διεθνείς μας εταίρους. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν περιφερειακής προστασίας και αλληλεγγύης θα αφορά την προστασία βέβαια, αλλά υπάρχει μέσα και μια πρωτοβουλία για ανάπτυξη από πλευράς της Ιορδανίας, και του Ιράκ που δεν θα έχει να κάνει μόνο με Σύριους πρόσφυγες αλλά και με άλλους πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες και από άλλους πληθυσμούς. Μετά από την έκκληση του κυριωτέρης προς, προς την Επιτροπή για τους πρόσφυγες, μιλάμε για 10.000 Σύριους στην Ευρώπη, για την επανεκατάσταση 10.000 που είναι η πιο ευάλωτοι στη Φιλανδία, την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, τις κάτω χώρες, την Ιρλανδία. Οι χώρες αυτές αποφάσισαν λοιπόν να δώσουν θέσεις μετεγκατάσταση ή ανθρωπιστική βοήθεια στους Σύριους αυτούς πρόσφυγες. Εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερα στις χώρες αυτές για την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν που συνεισφέρουν στη συλλογική μας βοήθεια επιπλέον και να ζητήσω από τις άλλες χώρες μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό. 50.000 Σύριοι ζήτησαν διεθνή προστασία στην Ευρώπη από την αρχή της κρίσης. 50.000 Σύριοι. Οι περισσότερες από τις αιτήσει αυτές έχουν κατατεθεί στη Σουηδία και στη Γερμανία. Οι Σύριοι πρόσφυγες ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές για να φτάσουν στην Ευρώπη ο δικός μέσω της Τουρκίας πρώτα απ' όλα, της Βουλγαρίας, της Ελλάδας ή τα Δυτικά Βαλκάνια. Ακολουθούν θαλάσσιες διαδρομές μέσω της Τουρκίας, της Αιγύπτου και το είδαμε με την τραγωδία αυτή της Λαμπεντούσα ότι προσπαθούν να πάνε και προς την Ιταλία. Διαπιστώνουμε ότι δίκτυα, εγκληματίες πολλές φορές εκμεταλλεύονται την απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πρόσφυγες αυτοί και τους εκμεταλλεύονται με το χειρότερο τρόπο. Η τραγωδία της Λαπεντούσα πριν από λίγες μέρες έδειξε κάποια πολύ σοβαρά πράγματα. Πρώτον, την στάση του Δήμου της Λαπεντούσα και του πληθυσμού της Λαπεντούσα που με αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα και τους ευχαριστούμε. Δεύτερον, κατέδειξε την αναγκαιότητα να αντιδράσουμε πιο αποτελεσματικά, χωρίς να εφησυχαζόμαστε, για να αντιμετωπίσουμε τα κλιματικά αυτά δίκτυα. Και τρίτον, κατέδειξε την ποιότητα και την διάσταση των ε, επιχειρήσεων διάσωσης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σεσίλια Μάλστρογ, μάλιστα αυτό ακριβώ πρότεινε στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων. Εννοείται ότι η ροή των προσφύγων αυτών προς την Ευρώπη δεν συγκρίνεται με τον αριθμό των προσφύγων οι οποίοι πηγαίνουν δίπλα στη Συρία, γύρω από τη Συρία. Οι άνθρωποι αυτοί οι απελπισμένοι που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη είναι όλο και περισσότεροι. Πράγμα το οποίο οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στα δικά μας εθνικά συστήματα. Στη Μάλτα, στην Κύπρο ή στην Ιταλία, όπως το είδαμε. Οι χώρες μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετόπου, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ελλάδα, όπου δεκάδες χιλιάδες καθημερινά φτάνουν στις χώρες αυτές, είναι περισσότερο εκτεθειμένες. Στην Ιταλία αυξήθηκε ο αριθμός με νέους πρόσφυγες οι οποίοι κατάφεραν να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι για τη δυνατότητα μεγαλύτερης ακόμα ροής προσφύγων. το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη όσον αφορά την, ε, τους πρόσφυγες, η Frontex με τα μέσα που έχει σήμερα στη διάθεσή της και μετά από διαβουλεύσεις με την ΥΠΑΤ αρμοστία του ΟΗΕ της Υπηρεσίας Μετανάστευσης την προηγούμενη εβδομάδα πήγανε στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η κατάσταση όπως την διαπιστώνουμε σήμερα δείχνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία μεταξύ μας. Δεν είναι ένα θέμα καθαρά εθνικό, είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα. Και η απάντηση αναμφίβολα δεν είναι να κλείσουμε τα εθνικά μας ε, σύνορα, να κλειστούμε, να οχυρωθούμε. Όχι. Η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη. Μια τέτοια κρίση μας επηρεάζει όλους και πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι με ένα πνεύμα μεγαλύτερης αλληλεγγύης. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, ήδη έχουμε ετοιμάσει μέτρα για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη με μια ενιαία προσέγγιση. Σε συνεργασία βέβαια πάντα με τον ΕΣΕΟ, με κονδύλια εκτάκτος για τους πρόσφυγες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέσω του Ταμείου για το Άσυλο και την Μετανάστευση. Η Frontex αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και στη Μεσόγειο και στο έδαφος και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες αυτές με μεγάλη υπευθυνότητα, γιατί όντως έχουν μεγάλη ευθύνη ώστε να διαχειριστούν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρώντας βέβαια και την αρχή της ε, μη, της μη επαναπρόθεσης με τα μέσα βέβαια που έχουμε στη διάθεσή μας τώρα απέναντι στην κρίση αυτή και στις ανάγκες τις σημερινές και τις αυριανές πρέπει να είμαστε σε θέση να βρούμε επιπλέον κονδύλια νομίζω ότι θα είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο η επιπλέον αυτή βοήθεια μπορεί να συμπληρωθεί και με επιπλέον δράση της ΙΖΙΟ και με επιπλέον ομάδες επίσης θα μπορούσαν να στηρίξουν τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και εφόσον επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση, κάτι το οποίο φοβόμαστε, αν χρειαστεί να έρθουμε αντιμέτωποι με ακόμα πιο μαζικές ροές προσφύγων, η Frontex θα πρέπει να μπορέσει να ενδυναμώσει τις κοινέ αυτές δράσεις της. Δεν θα είναι δυνατό κάτι τέτοιο χωρίς τα κράτη-μέλη να κάνουν επιπλέον προσπάθεια και να δώσουν επιπλέον χρήματα για να συντονιστούν οι δράσεις. Και όλα αυτά βέβαια μέσα στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Η υπηρεσία προστασίας των πολιτών πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο. Το 2006 είχαμε μιλήσει για τη δύναμη πολιτικής προστασίας και οι συνάδελφοι 3,5 χρόνια δούλεψαν σκληρά για να έχουμε μια απάντηση προληπτικά για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τα εθνικά μέσα σε προληπτικό επίπεδο. Δεν θέλουμε νέα μέσα, θέλουμε τα ίδια μέσα που έχουμε να τα οργανώσουμε καλύτερα ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κρίσεις, είτε είναι φυσικές καταστροφές, είτε είναι άλλες όπως αυτή τη φορά το θέμα των προσφύγων. Και έρχομαι και στο τελευταίο, κάτι πολύ ευαίσθητο που έχει να κάνει με τη Συριακή κρίση αλλά και άλλες κρίσεις στην περιοχή αυτή. Πρόκειται για την ε, τρομοκρατία, την απειλή της τρομοκρατίας και τους ε, ξένους οι οποίοι έρχονται, είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταξιδεύουν είτε στη Συρία είτε αλλού και είναι θύματα απαγωγών κλπ. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε όλοι αυτοί οι... που είναι θύματα ε, ποιον θύματα ακριβώ είναι. Δηλαδή αυτοί οι μαχητέ οι οποίοι πηγαίνουν, φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πηγαίνουν στι χώρε εκεί στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένω για να οδηγηθούν σε τρομοκρατικέ ενέργειε, δεν ξέρουμε ακριβώ το προφίλ του και πώ ακριβώ έχουν τα πράγματα εκεί. Αυτά λοιπόν. Η αλληλεγγύη είναι το πιο σημαντικό. Ανθρωπιστική βοήθεια απέναντι στη Συριακή κρίση και συγχρόνω όμω να είμαστε πολύ προσεκτικοί για του Ευρωπαίου πολίτε οι οποίοι στη Συρία και τι απειλή μπορεί να αποτελέσει κάτι τέτοιο για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα στοιχεία είχα να σας δώσω κύριε Πρόεδρε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της συναδέλφου Ζωζίεβα και Μάρστρομ. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς ε, κύριε Επίτροπε. Ξεκινάει λοιπόν τώρα η συζήτηση με τις δηλώσεις. Ε, ο πρώτος που έχει το λόγο είναι ο κύριος Βέιμπερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Αντιπρόεδρη, 93.000 νεκροί από τότε που ξέσπασε αυτός ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος στη Συρία αυτά λένε τα Ηνωμένα Έθνη. 2,6 εκατομμύρια πρόσφυγες εκτός ε, της ε, Συρίας, τόσα εκατομμύρια εντός της Συρίας, για να το ξεχνάμε. Και αυτό ο Λίβανος απαγόρευσε να κατασκευαστούν ε, νέοι καταπλησμοί προσφύγων, γιατί αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας του. Η Αίγυπτος και αυτή έχει προβλήματα, η Ορδανία και η Τουρκία βεβαίως προσφέρουν πάρα πολλά. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, η σύγκρουση που βιώνουμε στη Συρία η σύγκρουση αυτή είναι στην άμεση γειτονιά μας. Από την Κύπρο ουσιαστικά μπορούμε και να βλέπουμε το τι ακριβώς συμβαίνει στη Συρία. Γι' αυτό λοιπόν είναι σωστό που συζητάμε σήμερα το θέμα αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, για όλους μας ε, είναι σημαντικό να απευθυνθούμε καταρχήν στους ισχυρούς για να πάψουν αυτή την παράνοια και όσοι μπορούν να ασκήσουν επιρροή και σε αυτούς πρέπει να απευθυνθούμε. Αλλά πολύ συγκεκριμένα υπάρχει το πρόβλημα των προσφύγων. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν γιατί δουλεύει με αφοσίωση σε αυτό το θέμα για να σώσει ε, το πρόσωπο της Ευρώπης. Εμείς ως ΕΛΚ επιθυμούμε να παρακαλέσουμε το εξή. Αφενός η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει συγκεκριμένες ποσοστώσεις. Ακούγοντας τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, άκουσα μόνο λόγια, δεν άκουσα πράξεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, την σαφή έγκριση και από την υπατερμοστία των Ηνωμένων Εθνών ότι στην Ευρώπη πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ποσοστώσεις. Επ' αυτού είναι αρμόδια η υπατερμοστία. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να βοηθήσουμε επιτόπου στι όμορε χώρε. Ο επίτροπο, είπε έτσι λιγάκι συγκαλυμμένα ότι έχουμε προβλήματα χρηματοδότηση. Εγώ θέλω να το πω πιο ξεκάθαρα. Είναι ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση το ότι δεν υπάρχει ακόμα ο συμπληρωματικό προπολογισμό, ότι δεν είμαστε σε θέση ω Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβουμε τι ευθύνε μα. Το τρίτο που θέλω να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι λόγω των δραματικών εξελίξεων στην Λαμπεντούζα, λόγω αυτού παρά την το πρόβλημα της Συρίας πρέπει να προβαίνουμε σε διαχωρισμό ανάμεσα σε πολιτικά διοκόμενους και παράνομους μετανάστες. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Και το τελευταίο που θέλω να πω κύριε Πρόεδρε είναι ότι παρακαλώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συμπεριλάβει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξή του. Είναι προτεραιότητα. Δεν πρόκειται για τεχνικής φύσεως θέμα αλλά για το ε, τι πρόσωπο δείχνει τώρα η Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο συζητάει το θέμα αυτό και μάλιστα προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σουάμπαντα, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με ε, πρόσφυγες από τη Συρία. <clears throat> Μία από αυτές ήταν μία κυρία από την Παλαιστίνη που ανέφερε τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ως ε, Παλαιστίνια. Πρόσφατα πέθαναν πάνω από 100 άτομα στις ακτές έξω από τη Λαμπεδούσα που προσπαθώσαν να φτάσουν στην Ευρώπη. Είχαν όμως οι πρόσφυγες από την Παλαιστίνη προβλήματα για να μπορούν να έχουν ακόμα και προσωρινή άδεια κατάστασης διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπανε ότι πρωτού γυρίσουμε μπορείτε ίσως να μας δώσετε μια δυνατότητα να εκπαιδευτούμε, να έχουμε ορισμένε δεξιότητες. Δεν έχει νόημα όταν θέλουμε να έχουμε ειρήνη στη Συρία να είναι οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα είναι οι εμπειρογνώμονες για την ε, ανασυγκρότηση της χώρας μας. Εμείς θέλουμε να είμαστε οι εμπειρογνώμονες με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι, πρέπει να ανοίξουμε τα σύνορά μας για ένα περιορισμένο αριθμό προσφύγων, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και η Κομισιόν τόνισε ότι είναι διαφορετική κατάσταση σε διάφορες χώρες. Αν δείτε τα στοιχεία σε σχέση με τους πρόσφυγες, αν δείτε τον αριθμό των ετούντων ασύλου, και ιδίως αυτούς οι οποίοι αναγνωρίζονται ως έχονται στο δικαίωμα σε άσυλο. Βλέπετε μια τεράστια πολυπικίλια. Κάποιες χώρες κάνουν σωστά τη δουλειά τους, κάποιες άλλες χώρες όχι. Γι' αυτό κύριε Υπουργέ, εγώ απογοητεύτηκα τα μάλα από το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών. Άλλη μια μονάδα ειδική, μια task force. Θέλουμε δράση, δεν θέλουμε μονάδες μελέτης. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε ένα σαφές ψήφισμα για το τι θέλουμε να κάνουμε. Και συμφωνώ με τον κύριο Βέμπερ εγώ έκανα, έστειλα μια επιστολή στον κύριο Φαν Ρομπά, είπα θέστε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό δεν είναι μόνο ένα θέμα που απασχολεί του υπουργού εσωτερικών. Ξέρουμε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Είναι ένα θέμα για όλους μας, για όλη την Ευρώπη, για όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης, για όλους τους πρωθυπουργούς. Όλοι πρέπει να κάνουν τα απαραίτητα, τα απαιτούμενα. Ναι, πρέπει να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες. Αυτό δεν σημαίνει ότι απλώ του δίνουμε μια γωνιά να ζήσουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να κάποιες ε, δεξιότητες, να έχουν κάποια προσόντα, να μάθουν για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Θέλουμε μια Συρία χωρίς τον Ασάρτ και χωρίς τους τζιχαντιστές. Θέλουμε μια ελεύθερη και δημοκρατική Συρία. ζητήσαμε στο ψήφισμά μας τις χώρες που είναι όμορες της Συρίας. Παρακαλώ κρατήστε ανοιχτά τα σύνορά σας. Ιορδανία, Τουρκία, Λίβανος κτλ. Τα δικά μας σύνορα όμως είναι ανοιχτά. Τα σύνορα της Ευρώπης είναι ανοιχτά. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Θα πρέπει να σταθούμε ειλικρινείς. Γιατί δεν δημιουργούμε ασφαλείς ανθρωπιστικούς διαδρόμους για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Γιατί δεν δημιουργούμε εγκαταστάσεις προσωρινές διαμονής για τα άτομα αυτά για να τους βοηθήσουμε να έχουν κάποια εκπαίδευση και κατάρτιση. Θα πρέπει να σταματήσουμε τον ομό και σκληρό πόλεμο στη Συρία. Η καταστροφή των χημικών όπλων είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά όχι τίποτα παραπάνω από ένα πρώτο βήμα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας μέχρι ότου υπάρξει ειρήνη και συμφιλίωση στη Συρία. Και τότε θα γυρίσουν οι πρόσφυγες εκεί. Δεν θέλουν να φύγουν από τη χώρα του. δεν θέλουν να μείνουν έξω από τη χώρα του. Πρέπει όμω να του δώσουμε την ευκαιρία να οικοδομήσουμε μια νέα Συρία. Σε εργαστούμε λοιπόν μαζί του να καταπραίνουμε την τραγωδία τη προσφυγιά από του ανθρώπου, με το να του δώσουμε μια ευκαιρία να έχουν τη δυνατότητα να γυρίσουν στη χώρα του με τι κατάλληλε δεξιότητε, με την κατάλληλη παιδεία και να μεταλαμπαδεύσουν τη φιλοσοφία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Φερχόφ Στάτ. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή μπορούν να συμφωνήσουν με αυτό που προτείνει το Κοινοβούλιο που προτείνει να οργανώσουμε μία διάσκεψη ευρωπαϊκή για το θέμα αυτό. Αυτό ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του. Και θέλω να ακούσω πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή κατά πόσο το Συμβούλιο μπορεί να αναλάβει τη δέσμευση μαζί με την Επιτροπή να οργανώσουν τη διάσκεψη αυτή την ανθρωπιστική. Το είπανε και οι προλαλήσαντες ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο και δεν μπορεί να ζητάμε από τους άλλους να ανοίγουν τις πόρτες τους, τις χώρες τους, στους πρόσφυγες και να μην το κάνουμε εμείς. Η Γερμανία Προσωρινά θα δεχτεί 5.000. Η Σουηδία έχει δώσει επίσης ε, για 900 άδεια παραμονής. Η Φιλανδία κάνει μια αντίστοιχη προσπάθεια και τελεία. Άλλες χώρες δίνουν μια ποσόστοση για 50. Μα είναι σκανδαλώδες αυτό από μόνο του. Είναι κοινικό Συνεπώς, όσο γίνεται πιο γρήγορα να έχουμε τη διάσκεψη αυτή, όπου η Επιτροπή, το Συμβούλιο και όλες οι χώρες μέλη να καταλήξουν σε μια συμφωνία για το πώς θα μοιραστούν το βάρος της ε, κατάστασης αυτής. Δεν είναι δυνατόν μόνο η Σουηδία και η Γερμανία, πρέπει και άλλες χώρες να κάνουν ανάλογα κάποια προσπάθεια. Και έπειτα να βοηθήσουμε το Λίβανο και την Ιορδανία, γιατί τις χώρες αυτές πρέπει να τις βοηθήσουμε με κονδύλια και να τους δώσουμε και μια μακροοικονομική αρρωγή. Για τελειώσει οι χώρες αυτές δεν θα είναι πια σε θέση να αφήσουν τους πρόσφυγες αυτούς να μπαίνουν στις χώρες τους. Και τέλος, πρέπει να δούμε και το άλλο. Πρέπει ή δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί η οδηγία για την προσωρινή προστασία. Το ξέρετε και με το κοσυφοπέδιο. Ποια είναι η σωστή λύση, όπως είπε και ο κύριος Βόμποντα πολύ σωστά, οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να μείνουν για πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για προσωρινή προστασία μέχρι σε διεθνές επίπεδο να έχει λυθεί το ζήτημα αυτό. Οπότε η ερώτησή μου είναι πολύ συγκεκριμένη και σαφής κύριε Μπαρνιέ και προς τον Υπουργό της λιθανικής Κυβέρνησης. Είσαστε ε, διατεθειμένοι να οργανώσετε μια τέτοια ευρωπαϊκή ανθρωπιστική διάσκεψη. Αυτό ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε κι εμείς να συμμετέχουμε και πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να καλέσετε και τις γείτονες χώρες και τις Διεθνείς Υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και βέβαια εκπροσώπους από το Εθνικό Συμβούλιο της Συρίας και από άλλους που δραστηριοποιούνται επί τόπου. Τέλος, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου επαναλαμβάνοντας το εξής. Πιστεύω ότι η στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη Συριακή τραγωδία είναι μια ντροπή. Ναι, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των χημικών ε, όπλων. Ωραία, ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά οι σφαγές που γίνονται από το καθεστώς του Ασάτ, χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από χημικά όπλα, αλλά πάνω από 100.000 έχουν χάσει τη ζωή τους από άλλα μέσα και εμείς εξακολουθούμε να εθελοτυφλούμε στην τραγωδία αυτή. Σε 20 χρόνια. Στα βιβλία της ιστορίας θα μας περιγράφουν σαν δειλούς και ίσως να είμαστε πράγματι δειλοί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σαρτζεντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά ακούσαμε σήμερα. Δύο εκατομμύρια πρόσφυγες εκτός Συρίας, τέσσερα εκατομμύρια μέσα στη Συρία πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα, Τουρκία, Ιορδανία, Λίβανο, εκεί καταλήγουν οι πρόσφυγες. Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τίποτα, κλείνουμε το πορτοφόλι μας ή άντε το ανοίγουμε λιγάκι και δίνουμε κάποια μικρή βοήθεια, ενώ αφήνουμε την Τουρκία, το Λίβανο και την Ιορδανία μόνες τους να τα βγάλουν πόρα. Ε, όχι, νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε το πορτοφόλι μας καλά και να μην αρκεστούμε στα λίγα ψίχουλα που δίνουμε. Να μην διώχνουμε τους πρόσφυγες. Πρέπει να αφήσουμε 8.000 πρόσφυγες στις χώρες μας. Ο κύριος Φερχώστα θα αναφέρθηκε σε κάποιες χώρες οι οποίες κάνουν μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Η Σουηδία όντως είναι μια χώρα, αλλά υπάρχουν χώρες όπως και δικιά μου είπε 50 το 2013 θα υποδεχθεί. Ε, όντως είναι ντροπή. Οι περισσότερες ε, χώρες όμως στην Ευρώπη δεν κάνουν τίποτα. Το Βέλγιο για παράδειγμα. Η Λιθουανία επίσης. Και εδώ έχουμε υπουργό από τη Λιθουανία, ο οποίος μας ε, λέει τι θέλει να κάνει το Συμβούλιο και τι θα κάνει. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν για το πορτοφόλι, αλλά μια παραπάνω χειρονομία εσείς κύριε Υπουργέ πρέπει να μας πείτε εδώ ότι θα κάνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια η Λιθουανία. Και όχι μόνο για τους 50. Και οι υπόλοιπε 20 χώρες να έρθουν εδώ και να μας πούνε τι θα κάνουν. Και μόνο τότε θα έχουμε μιλήσει με ενωμένη φωνή και θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την Τουρκία και το Λίβανο και την Ιορδανία. Γιατί η μόνη λύση δεν είναι να ανοίγουμε το πορτοφόλι μας, πρέπει να δεχτούμε και τέτοιους πρόσφυγες στις χώρες μας. Η καταστροφή αυτή, η τραγωδία που είδαμε στη Λαμπετούσα πριν από λίγες μέρες, δυστυχώς ε, θα επαναληφθεί και θα τη βλέπουμε όλο και πιο συχνά από εδώ και πέρα. Όχι. Κάθε μέρα ξέρουμε ότι πνίγονται άνθρωποι στη Μεσόγειο. Η Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο πρέπει να ζητήσουμε και την βοήθεια των πρεσβειών. Και περιμένω τώρα, παρακαλώ, μια χειρονομία από την Λιθουανική Προεδρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο έχει το λόγο. Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει ένα κοινό σύστημα ασύλου. Αλλά πιστεύω όμω ότι αυτό το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί η ολέτρια ανθρωπιστική κρίση που λαμβάνει χώρα κοντά μα ο αριθμός των προσφύγων που εγκατέλειψαν ε, τη Συρία είναι ασύλληπτος και καθώς αυξάνεται ο αριθμός αυξάνονται και οι πιθανότητες οι άνθρωποι αυτοί να έρθουν στις ακτές μας. Είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι η αλληλεγγύη, συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη δεν πρέπει να είναι με τη μορφή εξαναγκασμού αλλά ε, μιας ηθικής επιταγής, κάτι που αναγνωρίστηκε και στην ε, συνάντηση της Γενέβης. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα πρώτα είναι να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, οι συζητήσεις μετά τη Λαμπεντουζά ελπίζω να προσφέρουν μάθημα. Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουμε περαιτέρω απώλεια ζώων είναι να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει με το να στουρθοκαμιλίζουμε και να ελπίζουμε το πρόβλημα να λυθεί από μόνο του. Αυτή η ανθρωπιστική κρίση δεν θα εξαφανιστεί από τα σύνορα της Ευρώπης ούτε απλά επειδή κλείνουμε τα μάτια. Δεν είναι πρόβλημα ούτε της Ιταλίας, ούτε της Ισπανίας, ούτε της Μάλτας και αυτό το αποδεικνύει ο αριθμός των ε, Συρίων προσφύγων ε, στη Γερμανία, στον Ρωμανό Βασίλειο και αλλού. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε περισσότερα, να αντιμετωπίσουμε την παράνομη εμπορία Σύριων ανθρώπων, είναι απελπισμένοι όταν έρχονται εδώ, να κάνουμε περισσότερα στη βοήθεια που στέλνουμε πιο αποτελεσματικά και πάνω απ' όλα να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τσίμα κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τον σεβασμό μου για τη στάση πολλών ανθρώπων στην ε, Λαμπεδούσα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι θα υποστούν ποινικέ κυρώσεις, βοηθήσαν άλλους ανθρώπους να σωθούν από τον πνιγμό. Υπάρχει η επίκριση λοιπόν που είναι απαραίτητη της Ιταλικής νομοθεσίας που κολλάζει τη βοήθεια που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι στους πρόσφυγες, αλλά πρέπει να τονίσω ότι και η στάση Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα όνειδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Εσωτερικών εν ώψη της κατάστασης της ε, ανθρωπιστικής καταστροφής της Λαπεντούσα και λαμβάνοντας υπόψη την συνυπευθυνότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα έσχος αυτό το οποίο έγινε. Το να μην αλλάζουμε τίποτα στο, στην ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και να λέμε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο δεν είναι μονάχα στουρθοκαμιλισμός, αλλά είναι απόλυτη ε, ανευθυνότητα από την πλευρά των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχεστε εσείς κύριε Βέμπερ από την Τσεσού. Έχετε μία θέση την οποία γνωρίζω ότι ακολουθεί και ο κύριος Φρίντεκ, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Ξέρετε πώς αντιμετωπίζει η Γερμανία τα θέματα αυτά. Αυτό για μένα είναι απόλυτα καταστροφικό. Είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχνάμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτοί που ζητούν άσυλο στη Γερμανία. Πιστεύω λοιπόν ότι εμείς θα πρέπει να οργανώσουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τη μετανάστευση και το άσυλο και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή της, κατάσ... της κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασύλου και τρίτον, θα πρέπει οι δυνατότητες που υπάρχουν ήδη σήμερα να ληφθούν υπόψη από τα κράτη-μέλη ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να βοηθήσουν τις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν ήδη ένα τεράστιο βάρος γιατί βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι δυνατό λοιπόν να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες και απλώς δεν πρέπει να συζητάμε περισσότερο, πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν και πάλι λίγη τουλάχιστον αξιοπιστία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αγωνίζεται για ένα αλληλέγγυο κόσμο και τέθη το θέμα του πώς οι άνθρωποι ε, εγκαθίστανται ως ετούντες άσυλο σε διάφορες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκρίνει τη Γερμανία με την Ιταλία, παραδείγματος χάρη. Αυτό δεν έχει καμία απολύτω σημασία, γιατί είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν καν σαν πρόσφυγε, αποθούνται σε χώρε όπω η Ελλάδα. Αν θέλουμε πραγματικά να κρατήσουμε ανοιχτά τα μάτια μα και να δούμε το πρόβλημα και να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε τέτοιε ανόητες συγκρίσει και να δούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση στη Συρία και έξω από τη Συρία, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια μεγαλύτερη αλληλεγγύη και πιο αποτελεσματική λειτουργία από εμά. Οτιδήποτε άλλο είναι ανάξιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Τσίμερα. Ο κύριος Σαλαβράκος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη αρχική φάση της επιχείρησης για την καταστροφή των χημικών όπλων έχει ήδη ξεκινήσει η παράδοση σε διεθνή έλεγχο και η καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της συρίας αποτελεί μια θετική εξέλιξη. είναι βέβαια σε εκτέλεση της συμφωνίας ή παρασουσίας. εγώ θα ήθελα να είχαμε την όχι και τόσο μεγάλη φαντασία την πρόταση πούτιν να την είχαμε κάνει εμείς για να δείξουμε ότι είμαστε εταίροι παγκόσμιοι σε επίπεδο κάπως υψηλό. ακολουθούμε και σε αυτή την περίπτωση παρότι σαν ευρωπαϊκή ένωση εμείς πληρώνουμε το μάρμαρο. ανησυχία ωστόσο μου προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με στοιχεία του οηε πάνω από δύο εκατομμύρια σύριοι έχουν εγκαταλείψει τώρα τη χώρα τους ενώ καθημερινά 8.000 άνθρωποι διασχίζουν τα σύνορα από ξηρά και θάλασσα. σημείωση στο σημείο αυτό. 10.000 ανθρώπους μόνο ε, έχουμε ήδη καλύψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 10.000 στα 2 εκατομμύρια. Είναι πολύ λίγο το ποσοστό. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερες δυνατότητες. Και δεύτερη σημείωση. Η Ελλάδα έχει 3 εκατομμύρια περίπου αυτή τη στιγμή μετανάστες. Όταν όλη η Ευρώπη για 10.000 συζητάει τόσο έντονα και τόσο πολύ και όλοι αποθούν την ιδέα. Έχουμε όμως το θάρρος εδώ στην ευρωπαϊκή ένωση να λέμε τους έλληνες των οποίων από τη μετανάστευση από αυτό το πρόβλημα όλες οι δομές έχουν καταποντιστεί να τους λέμε είτε τεμπέληδες είτε απατεώνες. από τη συνέχιση της εμφύλιας διαμάχης στη συρία με τις τραγικές συνέπειες στον άμαχο πληθυσμό υφίσταται κίνδυνος περιφερειακής διάχυσης της κρίσης. είναι απαραίτητο άμεσα να σταματήσει αυτή την κατάσταση και να βρεθεί πολιτική λύση. παρακαλώ να το βοηθήσουμε με εντονότερους ρυθμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ιμπατ Στάτλα θα ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις των ομάδων. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η τραγωδία στη Συρία είναι και το αποτέλεσμα λανθασμένης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Συρία. Άρα συνέβαλε και το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, Πολύ νωρίς εμείς ταχθήκαμε με την λεγόμενη Συριακή Αντιπολίτευση και ουσιαστικά ε, στηρίξαμε τρομοκρατικούς θυλάκους και αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα, οι θύλακοι αυτοί είναι συνυπεύθυνοι για δολοφονίες πολλών συμπεριλαμβανομένων και των χριστιανικών μειονοτήτων που ζουν στη Συρία. Εμείς στην Αυστρία έχουμε δεχτεί Σύριους πρόσφυγες και αν ακούσει τι λένε οι άνθρωποι αυτοί για αυτούς τους τρομοκράτες μισθοφόρους που εν μέρη χρηματοδοτούνται από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία και άλλες αραβικές χώρες ακούγοντας αυτές τις φρικαλές ιστορίες κατανοεί κανείς ότι δεν φταίει μόνο το Συριακό καθεστώς αλλά και αυτά τα δίκτυα τα οποία στην αρχή συγχρηματοδοτήθηκαν από τη Δύση. Ο πλούσιος αραβικός κόσμος, κυρίως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία με το υψηλότερο κατακεφαλή εισόδημα στον κόσμο, αυτοί φταίνε γιατί συγχρηματοδότησαν ε, τη Συριακή τραγωδία. Έστειλαν μισθοφόρους και φταίνε ε, διότι επίσης ε, χρηματοδότησαν και μεταφορά όπλων στους τρομοκράτες. Στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν έκαναν το ίδιο. Είναι λοιπόν συνυπεύθυνοι ως ε, αυτούργοι της ε, τραγωδίας και αυτό δεν έχει αναφερθεί στη συζήτηση και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πολύ ωραία. Ο Επίτροπος ε, παρακάλεσε σε ορισμένε ερωτήσεις να απαντήσει άμεσα. Κύριε Μπαρνιέ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρέμβω για λίγα λεπτά και να δώσω άμεσες απαντήσεις σε αυτό το στάδιο της συζήτησης, ιδίως στις εκκλήσεις πολλών από εσά, του κ. Βέμπερ, του κ. Σφόμποντα, του κ. Φερχόφστατ, της κ. Σατσεντίνη, της κ. Τσίμερ, του κ. Κίρκ Χοπ, που έθεξαν το θέμα αυτό των προσφύγων. Ανέφεραν ότι θέλουν να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή διάσταση για τα θέματα αυτά. Η απάντηση μου είναι ναι, εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, πιστεύω ότι μια τέτοια συνδιάσκεψη δεν θα είναι προσχρήσιμη θα είναι απαραίτητη αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε πολλά και πολλαπλά θέματα, για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα οποία δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε, να αντλήσουμε όλα αυτά τα διδάγματα αξιονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια και πώς να βοηθήσουμε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η πρώτη γραμμή και που δεν μπορούν να μείνουν μόνες για να αντιμετωπίσουν το θέμα της υποδοχής των προσφύγων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα ανηλεή αγώνα κατά των λαθρεμπόρων ανθρώπων με όλα τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει η θέση από κοινού των ε, εργαλείων πολιτικής προστασίας της χώρας μας. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό αν υπάρχει πολιτική θέληση και επίσης το θέμα της ανάπτυξης και της σταθερότητας των χωρών αυτών ώστε να μην χρειάζονται οι πολίτες τους να μεταναστεύουν προς την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι αρκετά σοβαρά θέματα ώστε να μπορέσουμε να <clears throat> ώστε να πρέπει να τα συζητήσουμε στο πιο υψηλό επίπεδο. Πρέπει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, οι, τα θεσμικά όργανα Τη Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την υψηλή αρμοστία, την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες να μπορέσουν να συζητήσουν για όλα αυτά τα θέματα. Thank. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για την σαφή απάντηση από την πλευρά της Κομισιόν. Θα ακολουθήσει και η αντίδραση φυσικά του Συμβουλίου. Ακολουθεί η κυρία Ματσιέ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε από την τραγωδία στη Λαμπαντούσα με τους πρόσφυγες που ερχόντουσαν από τη Συρία. Σήμερα φτάνουμε στο ημικύκλιο να συζητάμε και να σκεφτόμαστε τις μεταναστευτικές μας πολιτικές. Ο πόλεμος στη Συρία είναι καταστροφικός για όλους στη Συρία. Είναι χρέος μας λοιπόν να βοηθήσουμε το συριακό πληθυσμό και να του προσφέρουμε την αναγκαία προστασία. Τα Ηνωμένα Έθνη μιλούν για πάνω από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες, όπως είπε ο κύριος Μπαρνιέ. Η σύραξη όμως συνεχίζεται και θα φτάσουμε σε πάνω από 3 εκατομμύρια μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν τις γείτονες χώρες, οι οποίες με δίνουν πραγματική προστασία στους πρόσφυγες αυτούς, φροντίζοντας συγχρόνως να παραμείνουν κοντά στη χώρα τους. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές, οι οποίες 90% των προσφύγων έχουν στις χώρες τους και να αποδεσμεύσουμε κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συνεχίσουμε επίσης να αγωνιζόμαστε για την ειρήνη στη Συρία και για σταθερότητα στην περιοχή για όλους ε, αυτούς τους ανθρώπους. Όμως κύριε Επίτροπε, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούσαμε την απάντησή σας για τη διάσκεψη αυτή. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω εκ μέρους της δικιάς μας ομάδας, όπως και ο κύριος Βέμπερ νωρίτερα, οπότε πράγματι χαιρόμαστε πολύ που ανταποκρίνεστε θετικά στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αντιμετωπίζουμε και ένα πιο σφαιρικό πρόβλημα. Πώ να αντιμετωπίσουμε τι μεταναστευτικέ ροέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επίτροπο Μάλστρομ επίση ρωτήθηκε πώς και προσπαθεί να βρει λύση πώ να αντιμετωπίσουμε με περισσότερη αλληλεγγύη τις ροές αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν είναι έτοιμη σήμερα να απαντήσει στο αίτημα αυτό της Επιτρόπου Μάλστρομ. Είναι κρίμα. Ελπίζω η κυρία Μάλστρομ να μπορέσει κάποια στιγμή να εισακωστεί. Η κυρία Κιγιώμη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τι προτάσει που διατυπώθηκαν και την απάντηση του κυρίου Μπαρνιέ, εξ ονόμα της Κομισιόν. Είμαστε πολλοί που ζητούν κάτι τέτοιο, να υπάρχει μια επανεξέταση με συνολικό τρόπο των πολιτικών μετανάστευση και όχι μονάχα με ένα εμβαλωματικό και αποσπασματικό τρόπο. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική λύση στα διακυβευόμενα των μεταναστευτικών ρευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουν μεγάλη επίπτωση στην ευρωπαϊκό χώρο. Λοιπόν, άκουσα μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπε η Κομισιόν και περιμένω να ακούσω και την απάντηση του Συμβουλίου, ώστε για μια φορά το Συμβούλιο να απαντήσει όχι μονάχα σαν ένα αριθμητικό άθροισμα εθνικών πολιτικών, αλλά σαν μια συγκροτημένη πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα και τα προβλήματα που προκαλούν. Θα ήθελα να σταθώ εν τέλει και σε ένα τμήμα του ψηφίσματος αυτού σε σχέση με το άσυλο. Βέβαια πρέπει να υπάρξει κάποια βοήθεια στις χώρες οι οποίες είναι όμορες της Συρίας, αλλά πέραν αυτού θα πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει το δικό της τμήμα της, Ευρώπη, της ευθύνης σε ό,τι αφορά την υποδοχή των πληθυσμών αυτών που θέλουν να φύγουν από τη χώρα τους. Έχουμε με μεγάλη δυσκολία δημιουργήσει ένα καθεστώς για προστασία των προσφύγων, αλλά αν δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στην Ευρώπη με κάποια ασφάλεια, ή πρέπει να ακολουθήσουν διάβολους που είναι όλο και πιο πολυδάπανοι και τόσο όλο πιο επικίνδυνοι, αυτό δεν είναι λύση. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στα ρεύματα αυτά. Τα κάτι μελη έχουν ένα οπλοστάσιο μέτρων λειτουργικών, οικονομικών, θεσμικών για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν κανονικούς διάβλους εισόδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες θεωρήσει προξενικέ σε ανθρωπιστικό επίπεδο, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα επαναγκατάσταση και η Γαλλία έχει δεσμευτεί να κάνει και αυτή το δικό τη κομμάτι. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε μια πραγματική προσπάθεια αλληλεγγύη με του πρόσφυγε και τις χώρες που τους ε, υποδέχονται. Ευχαριστώ κυρία Βίξτρομ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ανθρωπιστική καταστροφή τεραστίων διαστάσεων στη Συρία. Ε, ο ανθρώπινος πόνος είναι διάχυτος και έχει φτάσει πια η στιγμή για μας στην Ευρώπη να καταδείξουμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Πρέπει λοιπόν όλοι στις χώρες μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Και αυτό μπορεί να γίνει μεταξύ άλλων εφόσον ε, καλέσουμε να έρθουν σε εμά ανθρώπους από τους καταβλισμούς στην Τουρκία, στην Ιορδανία και από αλλού, να τους καλέσουμε να έρθουν εδώ σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη η Σουηδία 10.100, ε, η Γερμανία πάνω από 5.000. Εάν λοιπόν και οι άλλες 26 χώρες ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, θα μπορέσουμε ήδη τώρα να προσφέρουμε προστασία σε περίπου 100.000 ανθρώπους. Βεβαίως το επόμενο βήμα είναι να οργανώσουμε αυτή τη σημαντική διάσκεψη για την οποία έγινε λόγος και πρέπει να μεριμνήσουμε πέρα από αυτό να προσφέρουμε και ε, ασφάλεια στους ανθρώπους προσφέροντάς τους ανθρωπιστική βοήθεια κυρίως σε αυτά τα προσωρινά προξενία που έχουν ανοίξει στους καταβλισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαρίστω να δώσω το λεπτό που έχω στη διάθεσή μου στον Υπουργό τη Λιθουανία, εάν έχει κάτι να μα πει. Γιατί εδώ που βρισκόμαστε, νομίζω ότι η δικιά σα σιωπή βαραίνει πάρα πολύ. Λέτε ότι χαίρεστε για τη συζήτηση αυτή που γίνεται κατεπηγόντω εδώ ότι το ψήφισμα σας ικανοποιεί, ναι, αλλά αναρωτιέμαι, το διαβάσατε το ψήφισμα αυτό. Και στη συνεδρίαση τη χθεσινή του Συμβουλίου οι Υπουργοί ασχολήθηκαν με τις προτάσεις μας στο Τζάκι αναρωτήθηκαν τι ανακοίνωση θα έπρεπε να έρθουν να μας κάνουν σήμερα στη συζήτηση αυτή κύριε Υπουργέ. Εγώ κατάλαβα ότι σημειώσατε την κατάσταση στη συνεδρίασή σας και ότι θα συζητήσετε στην επόμενη συνεδρίαση για το θέμα. Μα είναι έκτακτη η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ πραγματικά να λάβετε υπόψη σας το κατεπήγον της υπόθεσης. Όλοι οι συνάδελφοι που πήραν το λόγο πριν από μένα είπαν το ίδιο ότι χρειαζόμαστε εργαλεία, πολιτικές ικανότητες να δράσουμε τώρα αμέσως. Συνεπώς, εμείς αυτή την απάντηση θέλουμε να μας δώσετε. Σας παρακαλώ λοιπόν να πάρετε το λόγο και να πείτε το Συμβούλιο Υπουργών τι πιστεύει τελικά, τι θα κάνει. Ευχαριστώ λίγο ο Ο κύριος Φανέκη. Δεν είναι παρόν Ο Μποργέτσιο. Τρία σημεία θέλω να φέρω κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, πρέπει να ξεπεράσουμε τη συμφωνία του Δουβλίνου. Ε, να πηγαίνουν οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες. Ε, ανθίσατε η Γερμανία και να είναι ντροπή αυτό. Όσον αφορά τους ε, διακινητές ε, πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές ε, ποινές, να ξέρει ότι κινδυνεύει αυτός που συνέβη παραδείγματο χάρη είναι στην Λαμπεντούζα και στην, στο νησί την Τζίλια και είναι όλα ντροπή. Ευχαριστώ τον κύριο Μπαρνιά για αυτά που είπε για τις χώρες υποδοχής αλλά δεν ανέφερε την Ιταλία, την ξέχασε. Σήμερα ο πρόεδρος Μπαρόζο βρίσκεται στη Λαμπεντούζα και πρέπει να το ζητήσει αυτό από τον ε, Πρωθυπουργό Λέτα. Είναι ντροπή όπως λέει και ο Πάπας. Και θέλω επίσης από τον κύριο Μπαρόζο, επειδή είναι εκεί, να ε, επαληθεύσει, να διαπιστώσει κάτι γιατί δεν είναι ο στόχος να πάνε εκεί οι διάφοροι θύνοντες ε, να κάνουν κάποια διαφήμιση. Φαίνεται ότι τα πτώματα βρίσκονται σε μία αίθουσα τέσσερις ολόκληρες μέρες χωρίς κλιματισμό και παραμένουν εκεί τα πτώματα απλά και μόνο για να τα δείξουν στον κύριο Μπαρόζο και αυτό είναι ντροπή. Η κυρία Νέινσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Σήμερα μας απασχολεί το θέμα της αλληλεγγύης για, για τους πρόσφυγες. Αυτό είναι η λέξη κλειδί. Η τραγωδία που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες από τη Συρία είναι μια δοκιμασία για την έννοια της ελληνικής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υποδεχθούν πρόσφυγες και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και όχι μονάχα οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή το, οι κανονισμοί του Δουβλίνου 1 και 2 κάνουν υπεύθυνε για την υποδοχή των προσφύγων μόνο τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στο σημείο εισόδου των ε, προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτή η νομοθεσία. Υπάρχει πολύ διαφορετική ικανότητα υποδοχής στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Βουλγαρία δεν υπάρχει επαρκής ικανότητα υποδοχής προσφύγων. Πολλοί στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή θέλουν να κλείσουν τα σύνορα της Βουλγαρίας στους ε, πρόσφυγες. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση των χωρών της Μεσογείου που έχουν ξεπεράσει τις δυνατότητες υποδοχής τους. Θα πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν η απαραίτητη υποδομή ώστε οι πρόσφυγες παραμένουν κοντά στις αιστείες τους. Αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο σύνορο στην ε, Βουλγαρία είναι τα σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία. Η Βουλγαρία είναι μια χώρα η οποία υφίσταται μια τεράστια πίεση προσφύγων. Αυτό οδηγεί σε πολλούς κινδύνους για την εθνική μας ασφάλεια. Γι' αυτό κυρίε και κύριοι, σήμερα θα πρέπει να δώσουμε ένα σωστό μήνυμα και να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η κυρία Ντεκέιζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρώπη θέλει βέβαια να ανοίξει περισσότερο τα σύνορά της, δεν θα καταφέρει όμως να αποφύγει την ανθρωπιστική γενοκτονία που λαμβάνει η χώρα στην περιοχή, τώρα μάλιστα που πλησιάζει ο χειμώνας. Το κλειδί βρίσκεται στη Συρία. 6 εκατομμύρια μετατιζόμενοι μέσα στην ίδια τη χώρα. 2 εκατομμύρια στην γύρω περιοχή και 6.000 καθημερινά φτάνουν στο Λίβανο. Συνεπώς πρέπει να ασχοληθούμε πρώτα απ' όλα με το τι γίνεται εκεί και να κάνουμε διπλωματικές προσπάθειες. Είναι δύσκολο, είναι εφικτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνει ήδη. Πήγα στη Συρία και το Λίβανο πριν από 10 μέρες. Δεν ήξερα ότι ο πρέσβης μας στην ε, Δαμασκό λειτουργούσε με προσωπικό προσωπικό και ότι 10 μέρες το χρόνο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες ασφαλείας ε, ζει το προσωπικό. Ο Ντζενζίνε και η ομάδα του προσπαθούν να δράσουν απέναντι στην κυβέρνηση της Συρίας. Δεν ήξερα επίσης ότι οι διεθνείς μη ε, ε, κυβερνικές οργανώσεις και συνεργάζονται με την κυβέρνηση για να πάει ανθρωπιστική βοήθεια ότι διαφορετικές επαναστατικές ομάδες που μερικές φορές έχουν σχέση με την ε, Αλκαΐδα καθημερινά διαπραγματεύονται με τους διάφορους φορείς προκειμένου η βοήθεια να φτάσει εκεί όπου κατά χιλιάδες οι πολίτες βρίσκονται κλωβισμένοι. Και φυσικά υπάρχουν και οι βοήθειες της UNICEF, μια που χιλιάδες παιδιά δεν πάνε σχολείο εδώ και τόσα χρόνια. Χρειάζεται επιπλέον διπλωματική δουλειά. Η κυρία Γιώργε Βαχτές μου έλεγε ότι κατάφερε να πετύχει η θεώρηση και κάποιον από την ομάδα της για να μπορέσει να πάει να δουλέψει στη Συρία. Θέλω λοιπόν να ε, ποτισοφόρο τιμή στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ανθρωπιστική βοήθεια ζητώντας συγχρόνως να υπάρξουν και διπλωματικές ε, δραστηριότητες γιατί μόνο αυτές θα λύσουν το πρόβλημα στη Συρία. Ευχαριστώ. Κυρία Σάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και δυόμιση χρόνια είμαστε παθητικοί παρατηρητέ του πολέμου στη Συρία. Σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο περιθώριο. Όταν οι Σύριοι αντιμετωπίζουν τι χειρότερε ε, συνέπειε ενό πολέμου μέσω αντιπροσώπων που αποσταθεροποιεί όλη τη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει καμία προοπτική ε, λύση και καμία δυνατότητα να αποτρέψουμε μία δυνητική ανθρωπιστική καταστροφή με χρυσή όπλων μαζικής καταστροφής. Έχουμε χιλιάδες και εκατομμύρια πρόσφυγες και τεράστιες συνέπειες που προκύπτουν από αυτή τη μετακίνηση. Εμείς πρέπει να παίξουμε ένα πρωτοπόρο ρόλο στην ε, υποστήριξη σε ανθρωπιστικό επίπεδο και πράγματι θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τζόρτζεβα για τις προσπάθειές της για την ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει όμως να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκομένους για να υπάρξει μια λύση στα θέματα αυτά. Χαίρομαι λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διοργανώσει μια συνδιάσκεψη για να αντιμετωπίσει την έκκληση των ε, Ηνωμένων Εθνών. Μόνο ένα τρίτο των αναγκών έχουν καλυφθεί σε ό,τι αφορά τη στέγαση και την τροφή των προσφύγων. Θα πρέπει να σταματήσουν οι εσχρές συζητήσει όπως αυτές στην ε, Ολλανδία για το αν πρέπει να δεχτούμε 100 ή 150 πρόσφυγες στην χώρα μας όταν ο Λίβανος υποδέχεται πάνω από 6.000 κάθε μέρα. Έρχεται ο χειμώνας και δεν μπορούμε να αφήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να μένουν στην, στο ψύχος. Ευχαριστώ η κυρία Ντόμπς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ο αριθμός των προσφύγων που φεύγουν από τη Συρία για να ξεφύγουν από αυτό τον φρικαλαίο εμφύλιο πόλεμο είναι ανησυχητικός. Είναι αλήθεια ότι σήμερα το πρωί έχουμε στρέψει την προσοχή μας στο θέμα αυτό, αλλά είναι σημαντικό αυτοί που έχουν εκτοπιστεί από τη Συρία να προστατευτούν ικανοποιητικά από τη διεθνή κοινότητα και ενώ είναι σωστό να μην επέμβουμε στρατιωτικά, είναι επίσης σωστό να προσφέρουμε συντονισμένη ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ ιδιαίτερα γιατί υπάρχουν πολλοί που αντιμετωπίζουν ακόμα το φάσμα του θανάτου και της ε, λιμοκτονίας στη Συρία. Υπάρχουν οι χριστιανοί, είναι ο η μεγαλύτερη μειονότητα σε αυτή τη χώρα. Αναφέρονται δολοφονίες ε, που αφορούν αυτούς, ε, αναφέρεται φαίνεται ότι πολλοί τζιχαντιστές ε, προσπαθούν να τους ε, προσιλητήσουν ε, στο Ισλάμ και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Έτσι λοιπόν κύριε Επίτροπε απευθύνομαι σε εσά σε οποιαδήποτε συζήτηση και διάσκεψη που θα ακολουθήσει σας καλώ να προστατεύσετε τα θεμελιώδη δικαιώματα των χριστιανών στη Συρία και πρέπει να τους στηρίξετε με κάθε δυνατό μέσο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάδελφος Πίρκα, επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Ήδη έχουμε έναν που έχει χάσει από την κρίση στη Συρία και αυτός είναι ο λαός, οι πολίτες. Έξι εκατομμύρια πρόσφυγες στη χώρα και εκτός της χώρας. Αυτή είναι η συνέπεια. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι η πραγματική λύση μπορεί να είναι μόνο πολιτική. Και επ' αυτού έχουμε ήδη κάνει τα πρώτα βήματα και ελπίζω ότι αυτά θα καρποφορήσουν. Ε, αυτή τη στιγμή βέβαια πρέπει να καταφύγουμε σε βραχυπρόθεσμα μέτρα. Νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητα ε, τους καταβλισμούς, ε, να τους καταστήσουμε, να τους προσαρμόσουμε στο χειμώνα, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιβιώσουν ε, και συγκεκριμένα να παραμείνουν εκεί στην περιοχή. Το δεύτερο σημαντικό, και εδώ στηρίζω τα μέτρα της Επιτροπής, είναι ότι πρέπει επί τόπου, δηλαδή στα, στις περιοχές κοντά στα σύνορα της Συρίας, να τις στηρίξουμε τις περιοχές αυτές, να ιδρύσουμε σχολεία, γιατί ένας μεγάλος αριθμός των προσφύγων είναι για να εγκαταστήσουμε σύστημα ε, υδροδότησης ε, και άλλα μέτρα υποδομής γιατί πολλοί ε, παραμένουν εκεί. Επίσης το τρίτο πρέπει να επισημάνουμε στις αραβικές χώρες ότι δεν είναι δυνατόν ευθύνες να λαμβάνει μόνο η Ευρώπη και όχι οι όμορες χώρες οι αραβικές χώρες. Θα πρέπει και αυτές να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους ε, να δέχονται και αυτοί ε, πρόσφυγες ε, από τη Συρία. Εγώ μίλησα επιτόπου με πολλούς ανθρώπους και έκανα την εμπειρία ότι οι άνθρωποι αυτοί επιθυμούν να παραμείνουν στην περιοχή τους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει πρώτα απ' όλα υποστήριξη να προσφέρεται επιτόπου έτσι ώστε οι άνθρωποι μετά το τέλος της σύραξης να μπορούν το στομό δυνατόν να επιστρέψουν στη Συρία. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ψήφισμα για την Συριακή Σύρεξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προϋποθέτει μία έκκληση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει τις ευθύνες της να προστατεύσει το συριακό πληθυσμό. Γι' αυτό και ε, πρέπει να εκφράσει και αλληλεγγύη. Γι' αυτό λοιπόν κάνω έκκληση στην υπευθυνότητα των χωρών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν φτάνει μόνο οικονομικά να στηρίζουμε τις ε, χώρες που συνορεύουν με την Συρία. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Πρέπει να εξετάσει καλύτερα το κοινό σύστημα ασύλου. Να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 25 για τις θεωρήσεις, το οποίο επιτρέπει να δίνονται θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους. Να θέσει εφαρμογή το άρθρο 5 του Σέγγεν που επιτρέπει προσωρινά την πρόσβαση προσφύγων για ανθρωπιστικούς λόγους και να χρησιμοποιήσει επίσης πλήρως τα κονδύλια που έχει στην διάθεσή του για την επανακατάσταση, για το άσυλο και τη μετανάστευση και να χρησιμοποιηθούν επίσης τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας όσον αφορά όχι μόνο την προσωρινή διαμονή αλλά και τη μόνιμη διαμονή η Γερμανία και η Σουηδία προ το παρόν έχουν δεχτεί του περισσότερου πρόσφυγε, αλλά αυτό πρέπει να ισχύσει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο για τι χώρε αυτέ. Γιατί αλλιώ ε, δεν θα έχουμε τηρήσει την αρχή, την βασική, τη διεθνή που είναι τη μη επαναπρόθεση. Ευχαριστώ κύριε Γιαννάκου, έχει τώρα το λόγο. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Στη Συρία είναι προφανέ ότι γίνεται ένα βρώμικο πόλεμο ανάμεσα σε ένα δικτατορικό καθεστώ και σε ομάδε που θέλουν να εγκαταστήσουν δικτατορικό καθεστώ υπό το πρόσχημα μάλιστα τη θεοκρατία κύριε πρόεδρε αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι τέσσερα πράγματα πρώτα απ' όλα να πιέσουμε απόλυτα για πολιτική λύση μόνο πολιτική λύση μπορεί να δώσει την απάντηση δεύτερον να συνεχίσουμε την ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια στις όμορες χώρες με εποπτεία της ευρωπαϊκής επιτροπής επιτόπου κύριε πρόεδρε για να μην γίνει το αντικείμενο της ανθρωπιστικής βοήθειας αντικείμενο συναλλαγής των αντιμαχωμένων. τρίτον κύριε πρόεδρε είναι απόλυτη ανάγκη να γίνει αυτή η ευρωπαϊκή διάσκεψη στην οποία αναφέρθηκε και ο επίτροπος και τον συγχαίρω γι' αυτό και πρέπει να έχουμε και την απάντηση του συμβουλίου. από αυτή την ευρωπαϊκή διάσκεψη πρέπει να εξαχθούν και συμπεράσματα για τη γενικότερη μεταναστευτική μας πολιτική για τη γενικότερη πολιτική περί προσφύγων για το πώς κατανέμεται ανάμεσα στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης η ευθύνη. έχουμε παράδοση κυρίες και κύριοι στη βοήθεια προς τρίτες χώρες έχουμε παράδοση στην κάλυψη προσφύγων από όλο τον κόσμο αλλά η πολιτική μας παραπέει. πρέπει να υπάρξει μια συνεχής και συνεπής πολιτική που φυσικά δεν θα αποδίδει το βάρος με βάση τη συνθήκη δουβλίνο ii μόνο στις χώρες που βρίσκονται στη μεσόγειο αλλά θα το αποδίδει σε όλες τις χώρες και κυρίως κύριε πρόεδρε πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα και προς την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα και το δυτικό κόσμο ότι μόνο από κοινού και με απόλυτη πίεση μπορεί να υπάρχει ελπίδα για πολιτική λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έγγελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τρία σημεία θέλω να δείξω. Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι το άνοιγμα των συνόρων των χωρών κοντά στη Συρία ε, θα έχουν επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δίκιο. Και η Κύπρος και η Ελλάδα όμως είναι χώρες οι οποίες είναι γείτονες ουσιαστικά της Συρίας και δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς ενώπιον των μεσταναυτικών ρευμάτων. Όταν ζητούμε και σε χώρες όπως η Ορβανία ή ο Λίβανος να υποδεχθούν πρόσφυγες. Αυτό θα ήταν μια μορφή υποκρισίας από εμά. Δεύτερον είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο Επίτροπος κ. Μπαρνιέ, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει μια επανεγκατάσταση πολλών προσφύγων σε χώρες που έχουν τη δυνατότητα. Αλλά είναι πολύ λίγε οι χώρες, οι λεγόμενες μεγάλες χώρες μεταξύ αυτών που έχουν την θέληση να υποδεχτούν πρόσφυγε. Φαίνεται λοιπόν ότι η μεγαλοσύνη δεν έχει καμιά σχέση με το μέγεθος μιας χώρας. Μίλησε για την μη επαναπροώθηση ο κύριο Επίτροπο, γιατί αυτή η έννοια τη μη επαναπρόθεση ήδη αμφισβητείται από πολλού μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο. Τέλο, αναφέρθηκε σε ξένου μαχητέ ο κύριο Επίτροπο. Αυτό είναι και ένα κομβικό θέμα για το μέλλον. Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που από μέσα και από έξω από τη Συρία ε, παροτρύνουν αυτήν την ε, σύγκρουση και θέλουν να τη συνεχίσουμε. Ξέρουμε ότι είναι Πολλέ φορές εταίροι της Ευρώπης, χώρες όπως το Κατάρ που πρέπει να επανεξετάσουμε το ρόλο του. Θέλουμε να διαλυθεί η Συρία και τι θα κάνουμε με το μεταναστευτικό ρεύμα το οποίο θα προκύψει με μια τέτοια διάλυση της Συρίας. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να δώσουμε πολιτικές απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίλαν Μον έχει το λόγο. Τα νούμερα των προσφύγων από την Συρία είναι δύο εκατομμύρια σχεδόν και συγκεντρώνονται στην Ιορδανία, το Λίβανο, την Τουρκία και το Ιράκ κυρίω. Οι πρόσφυγες αυτοί καταδεικνύουν την τραγωδία που ζει η χώρα, όπω το λένε, το δείχνουν μάλλον και τα υψηλά νούμερα των θυμάτων. Πάνω από ένα εκατομμύριο είναι παιδιά, πάνε στι γείτονε χώρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, όπω είπε ο επίτροπο Ομπερνιέ, είναι ο πρώτο οδωρητής με ανθρωπιστική βοήθεια δηλαδή. Είπε επίση ο κύριος Μπαρνιέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση να αντιμετωπίσει το θέμα. Όμως, εκτός από την βοήθεια αυτή, πρέπει να προσπαθήσουμε να λύσουμε και την ουσία του προβλήματος, όσο γίνεται πιο γρήγορα, δηλαδή να σταματήσει η σύραξη. Μεγάλη βοήθεια προς τους πρόσφυγες, ναι. Αλλά πρέπει συγχρόνως να πείσουμε τους διεθνείς εταίρους αλλά και τις ε, αντιμεχόμενες δυνάμεις στη Συρία να καταλήξουν σε πολιτική λύση για να σταματήσει η σύραξη. Επιτέλους πρέπει να λάβει χώρα η διάσκεψη Γενέβη 2. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει αυτό τον Νοέμβριο. Τώρα, οι συνομιλίες ε, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για την καταστροφή των χημικών όπλων πρέπει να οδηγήσει και σε παρετέρω πρόοδο όσον αφορά την πολιτική λύση της σύραξης. Η πρόοδος για την καταστροφή των χημικών όπλων πρέπει όχι να επιβραδύνει, αλλά να επιταχύνει τη λύση του προβλήματος. Με βοήθεια λοιπόν προς τους πρόσφυγες, αλλά και τις χώρες που τους υποδέχονται και οι οποίες αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολη κατάσταση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά την Συριακή κρίση, εκεί κατορθώσαμε να αποτρέψουμε ένα ακόμα πιο τραγικό πόλεμο. Όμως ε, δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε αυτές τις ε, ροές μεταναστών και προσφύγων μάλλον που έχουν φτάσει σε πολλές χώρες μέσα Ανατολή αλλά και της Ευρώπης. Η πρόταση ψηφίσματος που συζητάμε είναι πολύ σημαντική και τη συμμεριζόμαστε, τη στηρίζουμε. Γιατί επιτέλους ε, επιβεβαιώνει κάτι που ισχύει στην περίπτωση της Συρίας και σήμερα πια επαναλαμβάνεται συνεχώς. Δηλαδή, Δηλαδή υπάρχουν ορισμένε χώρες ε, που έχουν προσπαθήσει περισσότερο στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Η Γερμανία δέχτηκε περίπου 15.000 αιτήσει, ε, η Σουηδία ε, και αυτή πάρα πολλές. Και έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό που προβλέπει το ψηφισμά μας, δηλαδή υπογραμμίζει ότι κατά την υποδοχή των προσφύγων από τη Συρία πρέπει να είμαστε περισσότερο συνοποιείς, να δείξουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα ε, κυρίως ε, απέναντι στα κράτη που δέχονται πίεση. Να υπάρχει μια ρήτρα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης γιατί είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαστε ένα συνονθήλευμα κρατών και αυτό αυτό χωρίς ε, καμία υποσημείωση. Πολλές χώρες, η Ελλάδα, η Μάλτα και άλλες ε, δέχονται συνεχώς ε, μεταναστευτικές ροές και αυτό το πρόβλημα δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν μόνες τους. Ο κύριος Στία έχει το λόγο. Πρόεδρε, πάνω από δύο εκατομμύρια πρόσφυγες και πάνω από 400.000 παιδιά ε, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Ε, χιλιάδες ε, είναι οι άστεγοι. Αυτά δεν είναι απλά στατιστικά δεδομένα, δεν είναι νούμερα, είναι ανθρώπινες ζωές. Πρέπει λοιπόν την Συριακή τραγωδία να τη συνδυάσουμε με την τραγωδία στη Λαμπεντούζα. Θα ήταν λάθος η συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική να μην λαμβάνει υπόψη όλε όλες αυτές τις εξελίξεις. Στη δική μου τη χώρα δεχθήκαμε πολλούς πρόσφυγες λόγω της επιθετικότητας του κυρίου Μιλόσεβιτς και ο πατέρας μου που ήταν ε, πρόσφυγας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μου έμαθε πάρα πολλά. Είναι πολύ σημαντικό για τους πρόσφυγες να μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αυτό πρέπει, εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Βεβαίως και στηρίζουμε το ψήφισμα, αλλά το κοινοβούλιο Συμβούλιο πρέπει να επικοινωνήσει περαιτέρω με εκείνες τις δημοκρατικές δυνάμεις στη Συριακή Αντιπολίτευση οι οποίοι προστατεύουν και όχι διώκουν τους χριστιανούς. Στόχος μας πρέπει να είναι ότι κάθε Σύριος πολίτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει στην πατρίδα του. Κυρία Σάγια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο και τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Πάνω από δύο εκατομμύρια πρόσφυγες προέρχονται από τη Συρία βρίσκονται στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στην Τουρκία κυρίω, Και αυτέ οι χώρε χρειάζονται οικονομική υποστήριξη και βοήθεια. Ο πρεσβευτή τη Ιορδανία μα είπε το καλοκαίρι ότι η κατάσταση γίνεται πραγματικά μια απειλή στην εσωτερική ασφάλεια της Ιορδανίας, πέραν της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν δεχτεί πρόσφυγες και αιτούμενους ασύλου, ιδίως γυναίκες και παιδιά η Γερμανία 5.000, η Σουηδία 900, η Φιλανδία 500. Αυτά είναι τα αριθμητικά στοιχεία που έχουμε για τις ποσοστώσεις που δέχονται οι χώρες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά οι ποσοστώσεις για τους πρόσφυγες είναι μονάχα ένα τμήμα της απάντησης. Χρειαζόμαστε την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Συρία. Χρειαζόμαστε να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία και να προστατεύσουμε τους πολίτες της χώρας αυτής. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η Προεδρεύουσα. Προχωρούμε με την οφθαρμοσυλληπτική και αγαπητοί συνάδελφοι, έχω λάβει 15 αιτήσει για ομιλία. Θα είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να ικανοποιήσουμε όλους. Θα δεχτώ μοναχά 7 ή 8 μιλητέ. <clears throat> και δίνω αρχικά το λόγο στην κυρία Σαροβιεύσκα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες της Συρίας, ο αριθμός των προσφύγων αυξάνει συνεχώς. Κάθε μέρα πάνω από 5.000 άτομα περνούν τα σύνορα της Συρίας. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό για τις χώρες της περιοχής οι οποίες υποδέχονται τους περισσότερους Σύριους πρόσφυγες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε τους ίδιους τους πρόσφυγες. Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την παράνομη μετανάστευση. Η Βουλγαρία διαμαρτύρεται για τεράστιες ροές Συρίων προσφύγων. Τρεις χιλιάδες μόνο έχουν πάνε, ενώ πολλές χιλιάδες έχουν ε, φτάσει στο Λίβανο. Δεν πρέπει λοιπόν να αποσταθροποιηθεί περισσότερο η περιοχή. Αντίθετα, μόνο 12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναλάβει δέσμευση και βοηθούν τους Σύρου πρόσφυγες. Μπορώ φυσικά να καταλάβω τις δημοσιονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές από τις χώρες αυτές, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες.

ότι αυτό που πρέπει να επιδείξουμε ως Ευρώπη είναι η ελεγγύη. Βλέπουμε ότι σε τελική ανάλυση δεν αλλάζει τίποτα στη Συρία, ακόμα και μετά από αυτά που είπε το Συμβούλιο Ασφαλείας για τα χημικά όπλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει την καθοδήγηση των διπλωματικών κινήσεων. Ευτυχώς βέβαια το ψήφισμά μας αναφέρει ότι αυτό το θέμα των προσφύγων είναι θέμα Ευρώπης και όχι μεμονωμένων κρατών που πλήττονται. Εγώ πιστεύω ότι είναι σωστή η πρόταση Μπαρνιέ να λάβει χώρα μια ε, ευρωπαϊκή ανθρωπιστική διάσκεψη. Είναι απολύτως απαραίτητο να μιλήσουμε όχι μόνο με τους ε, θεσμούς αλλά και με της ΜΚΟ και της ε, κοινωνίας ε, των πολιτών. Να υπάρξει ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα ασχοληθεί μόνο με το θέμα αυτό γιατί πρέπει να ληφθούν πολιτικά μέτρα αλλά και μέτρα έκτακτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Να αναθεωρήσουμε τη Συμφωνία Ντουβλίνο 2 όσον αφορά τη χορήγηση ασύλου γιατί εκεί δεν προβλέπεται η δυνατότητα να ζητήσει κανείς άσυλο σε άλλη χώρα πέρα από αυτή που έχει καταφτάσει. Ο ε, αυτό αφορά και την Ιταλία. Να προσφέρεται προσωρινή ανθρωπιστική διαμονή και ε, με τον τρόπο αυτό ας μην ξεχνάμε ότι θα αντιμετωπίσουμε την παράνομη διακίνηση ε, ατόμων γιατί αυτό είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας όπως προβλέπεται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Συνάδελφος Κέλλερ παρακαλώ έχετε το λόγο. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν ήδη να εγκαταλείψουν τη Συρία. Η Ευρώπη έχει δεχθεί περίπου 800.000 πρόσφυγες σε σύγκριση με 2 εκατομμύρια. Αυτό ε, δεν είναι τίποτα. Ε, πρέπει λοιπόν να αλλάξουν οι αριθμοί, να είναι πιο ξεκάθαροι. Όταν τα ε, όμορα κράτη της Συρίας λέμε πρέπει να, ανοίξουν, να κρατήσουν ανοιχτά τα σύνορα, ε, μάλλον εμείς πρέπει να ανοίξουμε και εμεί τα δικά μα και να προσφέρουμε τουλάχιστον μια ανθρωπιστική βίζα, μια θεώρηση ανθρωπιστική. Όχι συνεχώ να ψώνουμε τον δάχτυλο έναντι των άλλων, τώρα να δράσουμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε του ανθρώπου. δεν χρειάζεται να περιμένουμε την εντολή των ΗΠΑ. Τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένα για την κατάσταση αυτή, για πολλού ανθρώπου. Δεν πρέπει να μετακυλίουμε τι ευθύνε στα όμορα κράτη τη Συρίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Πάτη Αρμοστή για τους πρόσφυγες είπε ότι στη Συρία υπάρχει μια αιμορραγία γυναικών, παιδιών και ακόμα και άνδρων. Αυτή η μεταφορική παρουσίαση εξηγεί καλύτερα την κατάσταση εκεί. Πάνω από 2 εκατομμύρια έχουν φύγει από τη Συρία, πάνω από 4 εκατομμύρια υπάρχουν ως εσωτερικοί εκτοπισμένοι, προσπαθώντας να ξεφύγουν από ένα βίαιο πόλεμο όπου στο τέλος θα καταλήξουμε ο μισός πληθυσμό να, της Συρίας 10 εκατομμύρια ανθρώπων να χρειάζονται κάποιο είδους βοήθειας. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν υποστηρίζουν ούτε τον Ασάντ, ούτε τους, κατακαιρματισμένους, τους ηγέτες της κατακαιρματισμένης αντιπολίτευσης. Έχουμε όμως ενώπιόν μας μια υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ανοιχτές οι πόρτες για τα κράτη και πρέπει να παραμείνουν τα κράτη που είναι όμοιρα, όμορα της Συρίας, αλλά όχι τα ευρωπαϊκά σύνορα. Στρατιωτικοποιούμε τα σύνορά μας με τα αποτελέσματα τα τραγικά που έχουμε δώσει δίνουμε μονάχα μία βοήθεια 20 λεπτά του ευρώ ανά άτομο που είναι πρόσφυγας από τη Συρία. Χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια, χρειαζόμαστε επενδύσει για να δοθούν οι απαραίτητε υπηρεσίε, η στέγαση, η εκπαίδευση για όλου αυτού του πρόσφυγε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γκζιέμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μιλούμε εδώ για μια ανθρωπιστική καταστροφή στη Συρία. Τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο Ασφαλείας δηλαδή των Ηνωμένων Εθνών, καθυστερεί με την σύραξη αυτή. Πάνω από 100.000 Σύριοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Εκατομμύρια άλλοι έχουν μετατοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας και άλλοι εκτός των συνόρων της Συρίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από βοήθεια. Όμως πρέπει να βοηθήσουμε και τις θρησκευτικέ και άλλες μειονότητες που υποφέρουν από διώξεις και από τη βία στη Συρία, μεταξύ άλλων και οι χριστιανοί. Βλέπουμε επίσης τρομοκρατικές ομάδες μη συριακής προέλευσης που δρούν όμως στη Συρία και αποσταθεροποιούν την εσωτερική ασφάλεια στη χώρα. Δύο εκατομμύρια από βουλές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φτάνουν. Αυτό το έχουμε πει. Χρειάζεται μια πολιτική λύση. Οι Σύριοι χρειάζονται ειρήνη, κράτος δικαίου και το δικαίωμα να επιστρέψουν στις στέγες τους. Ευχαριστώ. What should be the priority? Ποια πρέπει να είναι η προτεραιότητα για τη Frontex και όλε τι άλλε ευρωπαϊκέ υπηρεσίε το να σώσουμε ζωές ή να, ζωές ή να αποθούμε του πρόσφυγε. Πού είναι η να αποθουμε του επιταγή για τον κύριο Μπαρόσο, ο οποίο βρίσκεται σήμερα ενώπιον των προσφύγων στην Λαπέδωσα. Τα περισσότερα κάτι έχουν αντιμετωπίσει το ρεύμα των προσφύγων με ένα αισχρότερο που χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική. Πρέπει να υπάρξει μια εστίαση πέραν αυτή για τα ανθρωπιστικά θέματα. Όλο και περισσότεροι πρόσφυγες όσο μένεται ο πόλεμο στη Συρία. Η, η Ευρώπη ζητά από τους ξένους, από τα ξένα κράτη να βοηθήσει του πρόσφυγε, αλλά η Ευρωπαϊκή ενώ δεν πρέπει να αφήσει την Συρία να αδειάσει από πολίτες. Πρέπει να υπάρξει μια αποτελεσματική βοήθεια μέσα στη Συρία. Αυτό σημαίνει μια πιο αποτελεσματική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία και στα άλλα σύνορα της Τουρκίας για να υποστηρίξει την ε, ε, υποδοχή των προσφύγων και να μην αφήσει να διαφθαρούν από των τζιχαντής. Πρέπει να ζητήσει επίσης και από την αντιπολίτευση στη Συρία να προετοιμάσει ένα δημοκρατικό μέλλον για τη Συρία. Κύριο Στογιάννοφ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το σημερινό μας θέμα είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπέρ των προσφύγων. Μα έχει ακούσει κάποιο από εσάς αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσει να αναφέρεται ένα συγκεκριμένο μέτρο. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Συζητάμε εντός, εκτός και επί τα αυτά για τα θέματα των ε, προσφύγων, ενώ έρχονται στη Βουλγαρία πρόσφυγες κάθε μέρα από την Τουρκία είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτείτε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι το κράτος μέλος το οποίο έχει δεχθεί το μεγαλύτερο αριθμό των προσφύγων. Το έχετε ξεχάσει. Η, Τουρ... η Βουλγαρία ήταν το τελευταίο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε αντικείμενο τρομοκραστικών ενεργειών από τους ε, Ισλαμιστές. Έχουμε λοιπόν τέτοια προβλήματα στην Τουρκία όταν εσείς μιλάτε για συνδιασκέψεις σε υποθετικό χρόνο. Συγχρόνως έχουμε ε, πρόσφυγες οι οποίες έρχονται στη Βουλγαρία και οι οποίοι πρέπει να, να συντηρηθούν με το τον κρατικό μας προϋπολογισμό. Λοιπόν, θα έπρεπε να κάνουμε μια σωστή ανέργεια για τα θέματα. Ο κύριος Λαντσπέργης έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο πόλεμος στη Συρία περιέχει στοιχεία τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί μετά τις επιθέσεις με αέρια του ίδιου του Σαντάμα απέναντι στο δικό του τον πληθυσμό. Τα χημικά όπλα είπαμε ότι πρέπει να καταστραφούν μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά δεν λέμε τίποτα για τους ίδιους τους δολοφόνους. ξέροντας τι επιπτώσεις υπάρχουν απέναντι στον πληθυσμό. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι ότι όλο και περισσότεροι οι Σύριοι πρόσφυγες φεύγουν προς πάσα κατεύθυνση στην Ευρώπη. Τίποτα δεν λέμε για το συριακό έγκλημα απέναντι στην ανθρωπότητα που μένει ατιμόρυτο. Για εγκλήματα πολέμου. Μόνο μιλάμε για την ροή των μεταναστών. δεν χρειαζόμαστε μόνο ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και ένα διεθνές δικαστήριο. Ευχαριστούμε. Τέλος, ο Ρίτσαρ Χάουιτ. Τρία πράγματα για τους, Συριανούς, για τους Σύριους πρόσφυγες. Πρώτον, δεν πιστεύουν στη διεθνή κοινότητα πια, γιατί λένε τους καταβλισμούς δεν έχουν πια ούτε τρόφιμα ούτε βοήθεια. Οπότε ε, λένε ότι αν υπήρχε ε, τέτοια βοήθεια και μπορούσαν θα επιστρέφανε στην ε, χώρα τους. Με κάθε σεβασμό όσον αφορά την κρίση στη Συρία ακούσαμε ότι χρειάζεται αλληλεγγύη. Και στους G20 ο Βρετανός Πρωθυπουργός τα είπε αυτά, αλλά δεν είναι από τις χώρες οι οποίες προσφέρουν βοήθεια στους πρόσφυγες. Το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι η παράνομη μετανάστευση στη Γαλλία είναι υπεύθυνη για την κατάσταση αυτή όταν πρόσφυγες μέσω Γαλλίας προσπάθησαν να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 60% της επαναγκατάστασης ε, γίνεται από δύο χώρες, μεταξύ των οποίων δεν είναι η δικιά μου. Υπάρχει κάποιο ηθικό δίδαγμα. Οι πρόσφυγες της Συρίας είναι απελπισμένοι το λόγο έχει τώρα ο Επίτροπος Μισελ Μπαρνιέ. Παρακαλώ, κύριε Μπαρνιέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι παρενέβησαν για το θέμα αυτό, για τις προτάσεις, για τις ιδέες που συνεισέφεραν, για το θέμα αυτό το οποίο είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Πέραν αυτών που είπα προηγουμένως, θα ήθελα όταν απείλησα για την έκκληση για μια συνδιάσκεψη για την αντιμετώπιση αυτών των ε, ανθρωπιστικών θεμάτων. Θα ήθελα να κάνω και μερικές περαιτέρω διευκρινήσεις και να δώσω μερικές συμπληρωματικές απαντήσεις. Η κυρία Σαρτζεντίνη αναφέρθηκε σε αριθμητικά στοιχεία. Μπορώ να σας δώσω αυτά τα οποία μας έρχονται από την αρμόδια διεθνή αρχή που είναι η ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες. Θέλω να σας πω ότι εδώ πρόκειται για μια αίτηση, ένα αίτημα προς τις ευρωπαϊκές χώρες να εξασφαλίσουν συνολικά 2.000 ε, εγκαταστάσεις προσφύγων και 10.000 ε, εισόδους προσφύγων. Και χαίρομαι γιατί μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δώσει μια θετική απάντηση και γι' αυτό θέλουμε να παρατηρούμε και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν και αυτές μια απάντηση, αν δεν το έχουν κάνει ακόμα. και αυτά έρχονται από τους φορείς που είναι σε θέση να ξέρουν καλύτερα ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Έρχομαι να απαντήσω τώρα σε αυτά που είπε ο κύριος Λόμπες Αγιλάρ. Σε σχέση με τις ανθρωπιστικές προξενικές θεωρήσεις. Εμείς θέλουμε να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή προσέγγιση για τα θέματα αυτά. Θέλω να σας υπενθυμίσω κύριε Αγγιλάρ όμως, ότι αυτό εναπόκειται στην κυριαρχικότητα κάθε κράτους μέλους να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι αυτό το εργαλείο της ανθρωπιστικής χορήγησης θεώρησης. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ιδέα αυτής της ανθρωπιστικης χορηγησης θεωρησης ειναι ενα ευαισθητο θεμα γι αυτο θεωρω οτι η ιδεα αυτή της συνδιασκεψης για την ανθρωπιστική δράση σε σχέση με τους πρόσφυγες θα είναι χρήσιμη, γιατί τα θέματα αυτά που είναι ευαίσθητα, αντί να είναι μονάχα η αποκλειστική υπόθεση κάθε χώρας, που γνωρίζουμε πόσο δύσκολη είναι και η εσωτερική πολιτική σε πολλά κράτη-μέλη με την ε, αναδίπλωση στο εσωτερικό της κάθε χώρας και την εθνική εθνικιστική στάση, θα ήταν πιο πρόσφορο να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση, μια ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε συνολικά τα θέματα αυτά και όχι ο καθένας να το κάνει μεμονωμένα. Ο κύριος Έγγελ, όπως κύριε Νένσκι, ανέφεραν ιδιαίτερες καταστάσεις χωρών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η Κύπρος, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ιταλία. Έχουμε αναπτύξει αποστολές συγκεκριμένες και την προηγούμενη εβδομάδα ακόμα για να μπορέσουμε με τις χώρες αυτές επιτόπου να ε, αξιολογήσουμε τις τεχνικές και οικονομικές ανάγκες για την υποδοχή των προσφύγων και επίσης είναι ορθό αυτό που είπε η κυρία Γιαννάκου και ο κύριος Σαλαβράκος σε σχέση με την Ελλάδα και την παροχή ασύλου από την Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει το σύστημα ασύλου και να μπορέσει για αυτό να πάρει και τεχνική βοήθεια και οικονομική από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Γιγιόμ ζήτησε περισσότερα χρήματα. Και εγώ το έχω τονίσει η κυρία Γιγιόμ. Σε ό,τι αφορά την ΕΚΟ, την ανθρωπιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πια άλλα χρήματα για το 2013. Έχουμε φτάσει τα όρια του τι μπορεί να πράξει η ΕΚΟ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το 2014 θα πρέπει να υπάρξει μια αντιμετώπιση μέσα στα πλαίσια των περιορισμών του προϋπολογισμού να απελευθερώσουμε περισσότερα κονδύλια για την ΕΚΟ και γι' αυτό τονίζω ότι αυτή η συνδιάσκεψη την οποία αναφέρατε θα έχει πολύ σημαντικό χαρακτήρα. Εν κατακλείδη θέλω ευχαριστήσω όλους και να αναφέρω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο είπε η κυρία ε, Ντεκέιζερ. Εγώ θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον πληθυσμό της ε, Λαμπεντούσα που έχει αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Δεν είναι μόνο αυτοί φυσικά, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι κάνουν ένα εξαίρετο έργο χωρίς να φαίνονται κατά ανάγκη πάντα και αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να τονίσω αυτά που κάνουν και οι υπάλληλοι των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Βηρητό, στην Δαμασκό. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε, όπως ελέγχθη, χρησιμοποιήσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την Συρία και μόνο 44% πηγαίνουν από αυτά τα κονδύλια στη Συρία, τα υπόλοιπα στι γειτονικέ περιοχέ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι αυτά πρέπει να περάσουν μονάχα από, μέσα από τι κρατικέ αρχέ που υπάρχουν ακόμα και από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Και αυτό θέλω να υπογραμμίσω το έργο των ΜΚΟ, γιατί πολλέ φορέ παίζουν και τη ζωή του οι άνθρωποι αυτοί. Θέλω λοιπόν εν κατακλείδη να πω ότι ενώπιον ενό τέτοιου δράματο που δεν αφορά μονάχα τη Σύρια αλλά κυρίω στη Συρία σήμερα, είναι απαραίτητο να δώσουμε μια κοινή απάντηση. Δεν μπορεί να είναι η εθνική αναδίπλωση η λύση και ο καθένα να κοιτάει μόνο την πάρτη του. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ευρωπαϊκό και επομένω θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό σε ευρωπαϊκή διάσταση, λαμβάνοντα υπόψη όλα τα εργαλεία που ανέφερα προηγουμένω που βρίσκονται στη διάθεσή μας, η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη για Ανθρωπιστική Βοήθεια, η θέση από κοινού των ικανοτήτων ε, υποδοχής, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η αναπτυξιακή βοήθεια, η υποδοχή των χωρών που είναι όμορες της Συρίας, άλλα θέματα της, ε, των συνθηκών υποδοχής των προσφύγων. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστούν στο κατάλληλο επίπεδο που είναι αυτό των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να λάβουμε υπόψη και την πολιτική διάσταση η οποία είναι πολύ σημαντική και αντικείμενο συζήτηση στι χώρε μα. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια ευρωπαϊκή πολιτική συζήτηση και όχι με μονομένε εθνικές συζητήσεις οι οποίε επικαλύπτονται. Σα ευχαριστώ λοιπόν για τι προτάσει και αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα λοιπόν, εκ μέρους του Συμβουλίου, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αναπληρωτή Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τον κύριο Λεσκεβίτσιτς. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητά μέλη. Είμαι ευγνώμων για την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη κάτω από αυτές τις συνθήκες οφείλουν να μεριμνήσουν για να αμβληνθεί ο πόνος στη Συρία. Και πράγμα ό,τι μπορούμε, δεν πρέπει όμως να ε, επαναπαυόμεθα στις ε, δάφνες μας ε, γιατί πάνω από δύο εκατομμύρια Σύριοι έχουν βιώσει τη δραματική εμπειρία του πρόσφυγα και άλλο 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα εγκαταλείψουν τη χώρα. Και δεν γνωρίζουμε και πόσοι άλλοι θα ακολουθήσουν το 2014. Βεβαίως, ο καλύτερος τρόπος ε, για να παρεμποδίσουμε την οδύνη αυτών των ανθρώπων είναι να εντοπίσουμε τα αίτια γιατί εγκαταλείπουν τη χώρα. Και το καλύτερο βέβαια θα ήταν μια, ε, η επίτευξη συμφωνίας ειρήνης διαρκείας. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι η Λιθουανική Προεδρία από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουμε ενεργά στην επίλυση του προβλήματος Συρίας. Τον προηγούμενο μήνα ε, προβήκαμε σε μία δήλωση ε, και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα μιας κοινή ε, ευρωπαϊκής ε, ενέργειας. Η Λιθουανική Προεδρία συνεχίζει τη συνεργασία με την ύπατη εκπρόσωπο και την αντιπρόεδρο της Επιτροπής και με άλλους άμεσα εμπλεκόμενους για να επανέλθει η σταθερότητα στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή. Συνεχίζονται βέβαια οι μάχες και κατόπιν τούτου πρέπει να καταφύγουμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε το σεβασμό του διεθνούς ε, ανθρωπιστικού δικαίου, την προστασία των αμάχων, μηδέν ανεκτικότητα απέναντι σε δολοφονίες, απαγωγές, μηδέν ανεκτικότητα απέναντι σε σεξουαλικά εγκλήματα και σε εγκλήματα με βάση το φύλλο ε, οι πιο ε, τρωτοί είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Όλοι λοιπόν οφείλουμε να μεριμνήσουμε για την προστασία των ανθρωπιστικά εργαζόμενων και του ετρικού προσωπικού. Να διασφαλίσουμε ε, ασφαλή, διάδρομο για να μπορούν να περνάνε τα φάρμακα και τα νοσοκομιακά αυτοκίνητα. Η Συρία οφείλει να ε, δώσει την άδεια για την ε, αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, να μπορεί να περνάει η βοήθεια αυτή μέσα στη Συρία και να μπορούν οι άνθρωποι να φεύγουν από τη Συρία μέσα από όλα τα δυνατά ε, κανάλια, όλες τις ε, διόδους. Τώρα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποστηρίξουμε την ανθρωπιστική βοήθεια, να συντονίσουμε τις προσπάθειες, να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της βοήθειας αυτής. Ε, νομίζω αυτό είναι καθοριστική σημασία για την κατάσταση, παρότι υπάρχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και περιορισμοί. Αν επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, τότε ε, ε, θα μειωθεί η αύξηση του αριθμού των προσφύγων περισσότερους από ό,τι προβλέπετε και ελπίζουμε κάποια στιγμή να αρχίσει να μειώνεται και ο αριθμός αυτός στο εγγύς μέλλον. Τώρα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση του κ. σχετικά με τον επάρξη ανθρωπιστική διάσκεψη, όπως αναφέρεται και στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Καλωσορίζω ανεπιφύλακτα την πρόταση και επιπλέον καλωσορίζω και τη θετική απάντηση που έδωσε ο Επίτροπος ε, κύριος Μπαρνιέ. Η Προεδρία είναι πρόθυμη να συνεργαστεί στενά επί του θέματος με την Επιτροπή, η οποία βέβαια φέρει τη βασική ευθύνη. Όμως μια διάσκεψη δεν αρκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίζει να συμπεριλαμβάνει τη Ρωσία και άλλους διεθνείς παίκτες ε, εμπλεκόμενους ε, στο θέμα της Συρίας. Αυτοί πρέπει να μοιραστούν μαζί μας τις ευθύνες και να προσπαθήσουν και αυτοί να λύσουν το ανθρωπιστικό πρόβλημα της Συρίας. Επιτρέψτε μου <clears throat> να δράξω την ευκαιρία για να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου προς τον κύριο Αγγιλάρ και αν θέλετε και στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ψήφισμα που καταθέσατε επίκαιρο και απαραίτητο όσο ποτέ. Πιστεύω ότι με τις κοινέ μας προσπάθειες θα καταλήξουμε σε μια κοινή στάση και θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Σύριους και θα επιφέρουμε ε, μακροπρόθεσμες λύσεις, μακράς διάρκειας. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Το Προεδρείο έχει λάβει μία πρόταση ψηφίσματος και η σχετική ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.30. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της ε, συναδέλφου Βεγνιό, αναγνώριση